Μέρα σας αγαπητή Επίτροπε, αγαπητή Σεσίλια. Άρχεται η σημερινή συνεδρίαση με πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη μια προφορική ερώτηση για τις διακρίσεις λόγω κάστας. Επιτροπή Ανάπτυξης είναι η επιτροπή που έχει καταθέσει αυτή την προφορική ερώτηση. Από ό,τι βλέπω όπως είναι λογικό άλλωστε, είναι η Εύα ε, Ζολή, η οποία έχει ως ε, συντάκτρια προφορικής ερώτησης πέντε λεπτά. Εύα, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε και είπατε πρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι, Απαρτχάιντ είναι ο όρος